σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο τη εμπορική και επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πρωτοβουλίες δημόσιου ιδιωτικού τομέα σε τρίτε χώρε. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την έκθεση που υιοθετήθηκε στην ίντα την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου με γραμματοτήσεις και των Επιτροπών ΙΜΚΟ και ΔΕΒΕ θέμα είναι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίκτυπός της στις πρωτοβουλίες δημοσίου ιδιωτικού τομέα, της ΣΔΙΤ. Ξέρουμε ότι πρόκειται για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για συνεργασία δηλαδή των δύο αυτών τομέων, για την παροχή σημαντικών υπηρεσιών, υπηρεσιών γενικού ε, ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, σε υποδομές, οδικές μεταφορές, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδροελεκτρικής ή ε, κοινωνικές υπηρεσίες, υγείας, ε, παιδείας και πρόσφατα είχαμε και ΣΤΙΤ στους τομείς των καινοτόμων ε, τομέων υψηλής τεχνολογίας. Δεν είναι κοινή πρακτική στις αναπτυγμένες χώρες περισσότερο χρησιμοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, ε, με συνεργασία δωρητών και τέτοιες ΔΙΤ είναι 15 με 20% του συνόλου των επενδύσεων σε τέτοιες αναπτυσσόμενες χώρες. Η έκθεση μου επικεντρώνεται κυρίως σε δύο βασικές προοπτικές των πρωτοβουλειών δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Η μία προοπτική είναι το ίδιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόθεση δηλαδή των εμπορικών μας συμφερόντων γιατί η συμμετοχή σε ΣΔΙΤ δίνει μεγάλη ευκαιρία σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ε, επεκταθούν σε νέες αγορές. Για παράδειγμα, με τις στις συνθήκες αγοράς, την σχετική ύφεση και την χαμηλή απασχόληση, ε, όλοι συμφωνούμε ότι χάρη στη ΣΔΙΤ και χάρη σε επέκτασή τους και σε άλλες ή ε, ε, διεθνείς ή με ευρωπαϊκές αγορές ή μόνο τότε οι επιχειρήσεις μας μπορούν να αναπτυχθούν και να έχουν μεγάλη επιτυχία και καλά αποτέλεσματα. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις μας να μπουν και να επεκταθούν και σε εξωτερικέ αγορέ, χρησιμοποιώντα χρησιμοποιώντας one-stop shop ή κοινέ πλατφόρμες και αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές ε, κάποιων θεσμικών οργάνων που ήδη συμμετέχουν σε τέτοια σχέδια, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχω όμω και αξιοποιωντα τι βελτιστες πρακτικε καποιων θεσμικων οργανων που ηδη συμμετεχουν σε τετοια σχεδια οπω ειναι η ευρωπαικη τραπεζα επενδυσεων εχω ομω και εναν αλλο στοχο που τον επιδιώκουμε στα πλαίσια τη αναπτυξιακή μα πολιτική που επίση είναι σημαντική. Μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειε ε, με τους στόχους μας, τους αναπτυξιακούς, προωθώντας τέτοιες ΣΔΙΤ. Για παραδείγμα, αναπτυξιακά προγράμματα υποδομών, ε, η πρόσβαση στο είδωρη στην ενέργεια σε αναπτυσσόμενε χώρε. Ένα σημαντικό τμήμα τη χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί οι ΣΔΙΤ πραγματικά θα μπορούσαν να, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Έχουμε βέβαια και κάποιε αρνητικές εμπειρίες, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι ΣΔΙΤ δεν σχεδιάστηκαν καλά, πήγαν στραβά ε, προσέκρουσαν σε υπερβολική γραφειοκρατία, σε κολυσιεργίες ή ε, καθυστερήσεις στη διαχείριση των προγραμμάτων. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Η εκθεσή μου πιστεύω ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να βελτιώσει την κατάσταση και επισημαίνω ότι η έκθεσή μου δεν συνιστά επουδενή απόπειρα νέας νομοθετικής πρότασης ή ενίσχυσης της γραφειοκρατίας. Όχι, επουδενή. Απλώς ε, παροτρύνουμε τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να στηριχθούν στις υπάρχουσες διατάξεις και να προωθήσουν τη συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιριών σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, η έκθεσή μου είναι ο καρπός αγαστής συνεργασίας ε, υπερκομματικής και συνεργασία μεταξύ πολιτικών ομάδων και επιτροπών και ευελπιστώ ότι θα υπερψηφιστεί και στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε 7 ομιλητέ για τη διαδικασία Catch the Eye. ξεκινούμε με τον κύριο Φραντζούλητσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, οι πρωτοβουλίε δημόσιου ιδιωτικού τομέα σε τρίτε χώρε ε, έχουν μεγάλη προοπτική για την αύξηση τη παραγωγικότητα και στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική θα πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει τι ευρωπαϊκέ εταιρείε στο εξωτερικό, όπου ακόμη αντιμετωπίζουν σημαντικού φραγμού στι συμβάσει του. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε διαγωνισμού και έχουμε κάνει κάποιε ε, προτάσει και για τη δημιουργία συμπράξεων και κοινοπραξιών. Θέλουμε να έχουμε ένα ε, σωστό θεμητό νομικό πλαίσιο που θα υποστηρίζεται καταλήλως. Πρέπει να δοθεί δυνατότητα στις διοικήσεις να ε, προετοιμάσει σωστά τις συμπράξεις και να έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει σε τέτοιες συμπράξεις σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει καταρχάς να επισημάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εφαρμόσει την αρχή της συνοχής στις πολιτικές εμπορίου, επένδυσης και ανάπτυξης. Όμως ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει τις αγορές δημοσίων συμβάσεων ανοιχτές στο διεθνή ανταγωνισμό, οι επιχειρήσεις της Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν φραγμούς στο εξωτερικό Απ' την άλλη πλευρά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης οφείλουν να εργάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές του οσα επιπλέον πρέπει να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες αρχές του οηε για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. επίσης οι αναπτυξιακές εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δημόσια αναπτυξιακή χρηματοδότηση δεν θα διοχετεύεται στις διάφορες πολυεθνικές αλλά θα χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των τοπικών οικονομικών δικτύων. τέλος εάν επιθυμεί η ευρωπαϊκή ένωση πραγματική ανάπτυξη και επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να υπάρξει διαγραφή των χρεών των αναπτυσσομένων χωρών έναντι του διεθνούς νομισματικού ταμείου της διεθνούς τράπεζας και της αφρικανικής ε, τράπεζας ανάπτυξης. Ο κύριος είναι αναφίβολο ότι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα ε, και καλέ συνέπειε, ιδιαίτερα για τις σύγχρονες υποδομές. Φυσικά έχουμε και κάποια αρνητικά παραδείγματα. Έχουμε κάποιες καταστάσεις ε, που πόρο απέχουν από το ιδεώδες. Ε, μερικές φορές όχι μόνο δεν έλυσαν προβλήματα, αλλά δημιούργησαν και προβλήματα. Γι' αυτό, κύριε Επίτροπε, παρακαλώ κοιτάξτε ένα πρόγραμμα που βρίσκεται στα ντουλάπια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά την Κροατία. Πρόκειται για μία οδική αρτηρία στην Ίστρα, στην Κροατία, που θα ήταν σημαντικό παράδειγμα συνεργασίας του ε, κροατικού δημοσίου και της γαλλικής επιχείρησης Μπουίκ. Γιατί να μην πραγματοποιηθεί αυτή η ΣΔΙΤ. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η οδική αρτηρία το Ι στην Ίστρα. Είναι κρίμα να βρίσκεται βλοκαρισμένη μια τόσο αξιόλογη πρωτοβουλία ιδιωτικού δημόσιου τομέα στα ντουλάπια της Ευρωπαϊκής, στα σιρτάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Βιέγκας, ε, η ΣΔΙΤ, οι πρωτοβουλία ιδιωτικού δημοσίου χαρακτήρα είναι μερικές φορές σύμπτωμα αυτού του ολοκληρωτικού καπιταλιστικού μοντέλου και αιτία της κρίσης του το μοντέλο αυτό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, δεν είναι το μοναδικό που θα πρέπει να υπάρχει, γιατί μερικές φορές ε, δεν αφήνει περιθώριο για επενδύσεις ε, και μάλιστα βρισκόμαστε στο έρμεο σημαντικών ομίλων και πολυεθνικών και για τις σημαντικές υποδομές αλλά και για την ενέργεια, την παιδεία ή την υγεία. Στην, ε, Πορτογαλία αυξάνονται οι ε, δαπάνες για τη ΔΙΤ ε, εις βάρος των κοινωνικών δαπανών. Δηλαδή ευημερία ναι, αλλά για λίγους μόνο, κυρίως για τις μεγάλες πολυεθνικές και τους ομίλους που καρπώνονται τα δημόσια κονδύλια. Αυτή, αυτό είναι το άνοιγμα που προτείνει και η Ευρώπη με το TTIP, που ουσιαστικά καταπολεμάει και διευρύνει ένα, ένα εργαλείο που είναι ουσιαστικά ο καρκίνος τη δημο, της, της δημοκρατίας μας. Στον τίτλο της έκθεσης, Πρόεδρε, ε, δηλαδή αυτού του είδους ε, ο αντίκτυπος, ε, θεώρησα ότι πρόκειται για αρνητικό αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο, στους πιο φτωχούς. Αυτούς δηλαδή λέμε να βοηθήσουμε και ταυτόχρονα τους ισοπεδώνουμε. Τελικά όμω εδώ πέρα, τελικά δεν πιστεύω ότι απλώ μιλούμε για τη σύμπραξη ιδιωτικού δημοσιοδομία. Πάντω η εμπειρία στη χώρα μα είναι ότι πολλέ φορέ δεν αποδίδει αυτή η σύμπραξη όπω το εθνικό μα σύστημα υγεία. Είδαμε ότι τελικά αυτό το που γίνεται είναι να έχουμε όλη την αναποτελεσματικότητα του δημοσίου και από την άλλη μεριά έχουμε ε, την ε, αδιφάγω κερδοσκοπία του ιδιωτικού τομέα. Επομένως ε, θα πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικό με αυτές τις ιδέες. Παρ' όλα αυτά πάντως, μπράβο στον εισηγητή γιατί αναγνωρίζει ότι πρόκειται για κάποιες αποφάσεις που θα πρέπει να είναι κυρίαρχες αποφάσεις των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ, Ροντρίγκης Πινέρα. Εκτός μικροφώνου. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τους σοσιαλδημοκράτες και πρώτα πρώτα σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά γιατί ήσασταν πάρα πολύ ε, δεκτικό σε συνεργασίες. Πάντως εμείς σοσιαλιστές θέλουμε να γίνει η μεταβολή της ε, νομοθεσίας τόσο ώστε να έχουμε λιγότερους κινδύνους από ε, αυτή την σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Δεν θα πρέπει ποτέ να επιλέγεται μια τέτοια συμπρασία διότι ωφελεί ε, την ε, διοίκηση γιατί δεν θα έχει ρίσκο να διαλέγεται γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να παρασχεθεί μια δημοσία κρατική υπηρεσία ε, στο χαμηλότερο κόστος και πιο αποτελεσματικά. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι ποτέ δεν θα θέλουν λύσουμε μια τέτοια σύμπραξη ούτως ώστε να ιδιωτικοποιηθούν τα, τα, τα κέρδη και από την άλλη μεριά να κοινωνικοποιηθούν αυτά που έχει κατακτήσει το δημόσιο. Οπότε γι' αυτό, αυτό που θέλουμε είναι ένα ξεκάθαρο και διάφορο το νομικό καθεστώς. Και επίσης έτσι να μπορούν να καλύπτονται τα έξοδα και οι πόροι του δημοσίου. Τελευταία κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ η, Ευρωπα... η Ευρώπη θα πρέπει να προσβλέπει στην ανάπτυξη ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών εντός των συνόρων της, αλλά και στου διεθνείς εταίρους τη. Η αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών θα πρέπει να είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες και ο βασικός τρόπος για να το πετύχουμε πέραν της υποχρεωτικής λογοδοσία κατά τη διαχείριση δημοσίων κονδυλίων είναι και η προώθηση ε, της ε, προσέλκυσης ιδιωτικού κεφαλαίου σε δημόσια σχέδια το αυξανόμενο εξωτερικό χρέος πολλών κρατών και η έλλειψη χρημάτων για υποδομές δημιουργούν περισσότερο χώρο για την εκλαΐκευση τέτοιων ΣΔΙΤ και εντός και εκτός της Ένωσης. Η εκλαΐκευση τέτοιων μοντέλων στις χώρες εταίρους θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να ενισχύσουν τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει με τρίτες χώρες να εξασφαλίσει ισότιμη μεταχείριση των επιχειρήσεών μας στις, στους δημόσιους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και ανοιχτή πρόσβαση τέτοιων συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ, Επίτροπος Χόγκαν. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Επίτροπο Βέλστρομ, Επίτροπο Εμπορίου απόψε. Ευχαριστώ τον εισηγητή κ. Ζαραντήλ και την Επιτροπή ΙΝΤΑ για τη δουλειά που έχουν κάνει για την έκθεση αυτή. Η έκθεση αυτή τονίζει τη μεγάλη σημασία των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που είναι εργαλείο για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αυτό έχει λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα ισχύσει και στι ε, γειτονικέ μα και αναπτυσσόμενε χώρε. Η έκθεση τονίζει την ευκαιρία που δίδεται από την Ευρωπαϊκή ε, Πολιτική Επενδύσεων σχετικά με τι ε, διαπραγματεύσει για επενδύσει σε τρίτε χώρε που ανοίγουν νέε αγορές για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Χαιρετίζουμε τις ε, προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια και για θεμητό ανταγωνισμό στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να διευκολύνονται ε, και να υπάρχουν στα αντίστοιχα κεφάλαια διεθνών συμφωνιών. Θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα θετικών προσπαθειών. Καταρχήν, ε, πρέπει να σας πω ότι ε, βελτιώνονται οι καινοτόμες λύσεις ε, και η καινοτόμος χρηματοδότηση που διευκολύνει έργα σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δεύτερον, η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να διευκολύνει την έρευνα και την ανάπτυξη προς όφελος του ανταγωνισμού δεν μπορούν να έχουν χώρο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τέλος οι συμπράξεις αυτές διευκολύνουν την πρόσβαση των εταιριών σε συμβάσεις με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να καλύπτεται το κενό όσον αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα των αγορών μεταξύ της Ευρώπης και άλλων χωρών. Και έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ευρωπαϊκών εταιριών σε άλλες χώρες. Η Επιτροπή ε, στην έκθεση θα ήθελε να αναφέρεται περισσότερο ε, ε, η δυνατότητα προστασίας επενδύσεων ευρωπαϊκών ε, ε, εταιριών σε τρίτες χώρες. Ιδίως σε περιπτώσεις ε, που υπάρχει θέμα επίλυσης σχετικών προβλημάτων. Θα συνεχίσει η Επιτροπή να ενισχύει τις προσπάθειές της ούτω ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Θα μεταφέρω τα σχόλιά σας στην Επίτροπο Μάλστρομ που είναι η αρμόδια Επίτροπος. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή εκ μέρους της. Ευχαριστώ. Κλείνει η συζήτηση.